Συνεδρίαση βάσει του άρθρου 56 και 57 του κανονισμού. Αναφέρθηκε, ζητήθηκε, μάλλον έγινε επίκληση του 56 57 του κανονισμού. είδαμε ότι δεν έγινε καμία προσφυγή βάσει του άρθρου 211 παράγραφος 4 του κανονισμού, άρα η ερμηνεία της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων στην συνάντησή της 14 Φεβρουαρίου του 2001 εγκρίνεται. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, των άρθρων 56 και 57, φεύγει από την ημερήσια διάταξη η έκθεση Ματιέ. Πρόκειται για ένα θέμα που συζητήθηκε επί μακρόν, τώρα υπάρχει μια σαφέστατη νομική εξήγηση. Η ημερήσια διάταξη τώρα, ας πούμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε καταρχά την δήλωση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την έκθεση προόδου 2010 σχετικά με την Κροατία. Συναντηθήκαμε χτες με τον Κροάτη Πρωθυπουργό, παρουσία και του κυρίου Σβόμποντα, και του Προέδρου της, ε, της αντιπροσωπείας με την Κορατία. Συζητήσαμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων της Κροατίας με την Ένωση και με μεγάλη ικανοποίηση σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να ε, παρουσιάσουμε το μέλλον της χώρας αυτής στο πλαίσιο αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία εδώ του Επιτρόπου κ. Φούλε και ζητώ από τον Προεδρεύοντα κ. Μαρτώνη να λάβει το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Γνωρίζουμε τη σημασία που δίδει η Ουγγαρία στο ζήτημα της ένταξης και σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο, κύριε Προεδρεόντα. Κύριε Μάρτονη. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνομαι στην Ολομέλεια με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά σήμερα. Η συνάντηση είναι μια επίκαιρη στιγμή για να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε την πρόοδο της ενταξιακής προοπτική της Κροατία και να παρουσιάσουμε τα σχέδια της Ουγγρική Προεδρία για το πρώτο αυτό εξάμενο του έτους. Καταρχά, θα ήθελα να καλωσορίσω την ενεργή εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης και την επικοδομητική συμβολή του στην γενικότερη συζήτηση για την διεύρυνση και την ενταξιακή πορεία της Κροατίας ιδιαίτερα. Όπως πολλές φορές υπογραμμίσαμε, η διεύρυνση ενισχύει την ειρήνη, την δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθά την Ένωση να πετύχει καλύτερα τους στόχους της πολιτικής της σε σημαντικούς τομείς που είναι βασικοί για την οικονομική ανάκαμψη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η διεύρυνση είναι βασική κατευθυντήρια γραμμή για την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση και προχωρά με ένα βήμα που καθορίζεται εν πολλής από την τήρηση από πλευρά των υποψηφίων χωρών των κριτηρίων της Κοπενχάγης και την ικανότητά τους να αναλάβουν τις ενταξιακές υποχρεώσεις. Η διεύρυνση είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού η δουλειά μας θα έχει ως στόχο να προωθήσει τις πολιτικές βάσει της συνένεσης ε, ε, που υπάρχει σχετικά με την διεύρυνση και που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2006 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου του 2010, που υποστηρίχθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά την Κροατία, η ολοκλήρωση των μεταξιακών διαπραγματεύσεων όπως αναφέρουν και τα συμπέρασματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πολύ κοντά μας. Ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Υπό τον όρο βεβαίω ότι η Κροατία θα καλύψει τα υπόλοιπα ορόσημα για να κλείσει τα διαπραγματευτικά κεφάλαια. Επίσης, θέλουμε να ολοκληρωθεί η σύναψη της συνθήκης προσχώρησης και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για προσχώρηση της κρατίας στην Ένωση, κάτι προς το οποίο προσβλέπουμε. Όπως υπογρανίστηκε λοιπόν στο ψήφισμα σας, το εξάμεινο αυτό θα είναι κρίσιμο για, την, για τις διαπραγματεύσεις της χώρας αυτής. Θα ήθελα να μιλήσω εντάχει για τα κρεμή ζητήματα. Μέχρι τώρα και από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων 33 από τα 35, 34 από τα 35 διορθώνει ο κεφάλαια έχουν ξεκινήσει για τις διαπραγματεύσεις. Από αυτά 28 έχουν κλείσει προσωρινά. Άρα είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, πρέπει να κλείσουν κανένα δυο δύσκολα κεφάλαια όπως ο ανταγωνισμός, η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου, η αλληλεία, η περιφερειακή πολιτική και ο συντονισμός των διαθροντικών εργαλείων, το δικαστικό και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και τα δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Κάποια από αυτά έχουν και δημοσιονομικές συνέπειες βεβαίως. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την τια που υιοθετήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο υπογραμμίσαμε βασικά θέματα που απαιτούν περαιτέρω δουλειά στου τομεί αυτούς. Τα γνωρίζετε. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ωστόσο κάποια σημεία που αντικατοπτρίζονται και σωστά στο ψήφισμά σα. Άλλωστε, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η Κροτία κατέβαλε σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς μεταξύ των οποίων το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι χρειάζονται και περαιτέρω προσπάθειες. Τούτο αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και την αποτελεσματικότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο. Επίσης το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Κροατία να προωθήσει τις προσπάθειές για να καλύψει τα υπόλοιπα ορόσημα όπως την προετοιμασία ε, πιστικών αποτελεσμάτων, ιδίως στην πολιτική ανταγωνισμού και τα ζητήματα της δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να υπογραμμίσω εδώ τη σπουδαιότητα που δίνουμε στη διαδικασία παρακολούθησης για την προσαρμογή και υλοποίηση του κεκτημένου, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί η διοικητική ικανότητα και να υπάρξει επαρκές και πιστικό ε, ιστορικό. Η αξιολόγηση της Επιτροπής στην πρόοδο στον τομέα της δικαστικής εξουσίας και των ε, δεμελωδών δικαιωμάτων το Μάρτιο θα είναι πολύ σημαντικό ορόσημο για το ενδεχόμενο του, της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 23 αργότερα μέσα στο εξάμεινο. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το Διεθνέ ε, Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία, το Συμβούλιο διαπίστωσε εν γέννη την καλή συνεργασία τη ε, Κροατία με το δικαστήριο, επαναλαμβάνοντα ωστόσο ότι είναι αναγκαία η πλήρη συνεργασία. Αυτό ευθυγραμμίζεται άλλωστε και με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Τώρα που ξεκίνησε να εξετάζει νέα στοιχεία η σχετική task force, το Συμβούλιο ζήτησε από την Κροτία να συνεχίσει τις διοικητικές έρευνες για να παρασχεί τα ελείποντα στρατιωτικά έγγραφα. Επιπλέον το Συμβούλιο Υπογράμισε τον ενεργό ρόλο της Προεδρίας στην περιφερειακή συνεργασία και τη βελτίωση των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες καθώς και τις προσπάθειές της που έχουν ως στόχο τη συμφιλίωση ε, των λαών στην περιοχή. Η συμφωνία, υπογραμμίστηκε η συμφωνία διαιτησίας ε, με την Σλοβενία τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι που θεωρούμε πολύ ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα. Λαμβάνοντα υπόψη τη σπουδαιότητα των καλών γειτονικών σχέσεων, το Συμβούλιο ενθάρρυνε την Κροατία να εκμεταλλευτεί την πρόοδο αυτή στις προσπάθειές της για την επίλυση όλων των εκκρεμών διμερών προβλημάτων και ζητημάτων συνεργασία με τις εμπλεκόμενες χώρες. Συμπερασματικά, θέλω να επαναλάβω ότι πολλά ακόμα παραμένουν να γίνουν κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας η Κροατία, η Κροατία θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καλύψει τα υπόλοιπα ορόσημα, να διαφυλάξει και να βελτιώσει ό,τι έχει ήδη επιτευχθεί και να ολοκληρώσει και να καλύψει όλες τις άλλες υποχρεώσεις που είναι ακόμα εκκρεμείς βάσει και των διαπραγματευτικών ορισίων. Από πλευρά μας είναι αυτονόητο ότι θέλουμε και επιδιώκουμε την υποστήριξη και συνεργασία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως πρώτα απ' όλα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η χρονική στιγμή για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις επιτυχώς όπως υπογραμμίστηκε που όπως υπογραμμίστηκε αποτελεί προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας να ολοκληρωθούν λοιπόν αυτά μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Προεδρεύοντα. Η πολιτική γειτονία πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιοχή της Μεσογείου, η εταιρική σχέση προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πρώτα και κύρια θέματα, ωστόσο τα θέματα των Βαλκανίων. Ο κύριος Επίτροπος ο Στέπαν Φιούλα είναι αρμόδιος για αυτή την πολιτική γειτονία. και για την διεύρυνση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισήγητη για την Κροατία, τον κύριο Χάνες Σβόμποντα και να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ισοδίκαια προσέγγιση και μια ισορροπημένη έκθεση. Αναγνωρίζεται η εντυπωσιακή πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την Κροατία στο να ανταποκριθεί στα κριτήρια για την ένταξη, αναγνωρίζοντας ωστόσο επίσης τις προσπάθειες που είναι αναγκαίες επίσης για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία προσωρινά έχουν κλείσει 28 <clears throat> από τα 35 κεφάλαια υποδιαπραγμάτευση η υπουργική διάσκεψη της 19ης Απριλίου θα έπρεπε να είναι σε θέση να κλείσει και πρόσθετα κεφάλαια που θα έχει είτε υλοποιήσει είτε θα βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση των οροσίμων η Κροατία. Και όπως σημειώθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2010, είναι στο χέρι μας να πετύχουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Όπως με όλες τις διαπραγματεύσεις, τα πιο δύσκολα θέματα απομένουν ακόμα στην τελική ε, φάση αυτή. Και όπως ο Υπουργός, ο Προεδρεύων της ε, Ουγγρικής Προεδρίας ανέφερε προηγούμενα, έχει αναφέρει τον στόχο της η Ουγγρική Προεδρία να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις κατά το πρώτο ήμιση του 2011 εφόσον θα υλοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, και τα ε, ε, τα ορόσημα. Είναι σημαντικό αυτό να συνεχίσει η Κροατία να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τα όσα απομένουν έγκαιρα. Οι κύριες απομένουσες προκλήσεις είναι τα θέματα για το κεφάλαιο 23 τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κεφάλαιο 8 για την πολιτική για τον ανταγωνισμό. Η Κροατία εργάστηκε σκληρά, εργαζόταν και εργάζεται σκληρά για αυτά τα δύο παιδεία. Τώρα όμως ήρθε η χρονική στιγμή να περάσουμε στην τελική ευθεία. Όσον αφορά το δικαστικό και τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι τα κύρια θέματα που καλείται η Κροατία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Και αυτά είναι να θεσπιστεί μια αξιόπιστη <clears throat> προσπάθεια στην καταπολέμηση της διαφθοράς η ενδυνάμωση της λογοδοσίας ε, της αμεροληψίας ε, όσον αφορά αυτό το σκέλος ε, και την επαγγελματική αποδοτικότητα του δικαστικού σκέλους να αντιμετωπιστεί το θέμα της ατιμορρησίας των εγκληματιών πολέμου και να υπάρξουν και προγράμματα για την επιστροφή προσφύγων, βελτιώνοντας την υλοποίηση των δικαιωμάτων για τις μειονότητες. Πλήρης συνεργασία. Αυτό εξακολουθεί και απομένει ως ε, απέτηση έναντι της Κροατίας. Σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς ε, σαφή ορόσημα πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από την Κροατία για κάθε ένα από αυτά τα ορόσημα και απαιτήσει και θα αναφερθούμε σε έκθεση, στην προσωρινή μας έκθεση για αυτά τα θέματα αυτών των κεφαλαίων μέχρι τα μέσα Μαρτίου ακούσαμε και είχαμε μια πολύ σημαντική ε, επικοδομητική συνάντηση ε, σε σχέση με την χθεσινή έκθεση. Συζητήσαμε το θέμα του να διατηρηθεί η προώθηση των διαπραγματεύσεων και να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα εναπομείναντα θέματα. Οι κροατικές αρχές έχουν καλό συνειδητοποιήσει αυτά τα οποία πρέπει ακόμα να πράξουν. Πράγματι, με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα ότι με διασφάλισαν από πλευράς των προσωπικών ε, δεσμεύσεων της Πρωθυπουργού ότι θα συνεχιστεί με πλήρη ταχύτητα αυτή η προσπάθεια μέχρι ότου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με εκείνους που ζητούν να αντιμετωπιστεί το θέμα της Κροατίας χωρίς ε, οποιασδήποτε εκτόσεις ε, ή επαναχωρήσεις. Οι αρχές ε, των, του πλήρους σεβασμού των υποχρεώσεων που πρέπει να υλοποιούν τα υποψήφια κράτη και ο πλήρης σεβασμός των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απομένουν τα ορόσημα της διαδικασίας διεύρυνσης. Αυτή είναι η πεντουσία της αξιοπιστίας αυτής της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να δίνει πλήρη υποστήριξη προς την Κροατία, που εργάζεται σκληρά να επιτελέσει τους στόχους της της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιος και εδώ ακολουθώ την γραμμή του κύριου Μάκλονη ότι τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη μπορούν να ολοκληρωθούν. Μόλις θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των υπολείπων ακόμα ανοιχτών κεφαλαίων. Και είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο <clears throat> όταν θα ζητηθεί να υποβάλει την γνωμοδότησή του θα το κάνει και θα διαδραματίσει αυτό το σημαντικό ρόλο σύμφωνα με την πολύ επικοδομητική προσέγγιση που είχε υιοθετήσει και που είχε δείξει για την συνολική διαδικασία της ένταξης της Κροατίας. Από με τον εισηγητή σας κύριο Σβόμποντα πιστεύω ότι οι πολίτες της Κροατίας αφού ζητήθηκε να υιοθετήσουν τους στόχους της ένταξης της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση στο δημοψήφισμα να, μετά από το δημοψήφισμα να εκλέξουν τους εκπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Χάνες Φόμποντα, ο εισηγητής και αντιπρόεδρος Παρακαλώ, από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές και εισηγήτριες για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και που οδήγησε στο ότι ελπίζω να έχουμε μια έκθεση που θα βρει ευρεία συνένεση και έγκριση. Θέλω να ξεκινήσω κύριε Πρόεδρε με την σίγουρα πολύ επιτυχή επίσκεψη της Πρωθυπουργού ε, της Κροατίας εδώ στο σώμα μας. Εσείς επισημάνατε Πρόεδρε ότι δεν είναι μόνο σημαντική ένταξη της Κροατίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ίδια την Κροατία αλλά ως μήνυμα προ τα κράτη της ε, περιοχής αυτής. Και για τις μεταρρυθμίσεις. Όταν κάνει τη δουλειά, τη δουλειά της μια χώρα πρέπει να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και να δοθεί η ιδιότητα κράτους μέλους σε αυτή τη χώρα. Και όπως ανέφερε και ο Προεδρεύων κύριος Μάτβονη και ο κύριος Επίτροπος δεν έχουν όλα ακόμα ολοκληρωθεί. Πρέπει ακόμα να γίνουν τα τελευταία για τις μεταρρυθμίσεις ώστε να φτάσουμε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο και να μπορέσει να υπογραφεί η συμφωνία της ένταξης. Και σε σχέση με το ότι με την αντιπαράθεση στον κόλπο του Μπεράντ με την Σλοβανία θα πρέπει να εξευρεθεί μια διαδικασία για την επίλυση αυτού του επίμαχου θέματος και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για παράδειγμα για όλη την περιοχή και για το Κωσυφοπέδιο να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις αλλά μέσω διαβουλεύσεων να επιλύονται τα προβλήματα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι πρέπει να πορευτούν προς μία ενιαία κατεύθυνση. Συμπολίτευση, κυβέρνηση δηλαδή και αντιπολίτευση. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις ε, ειδήσεις μας. Συζητήσαμε και τα θέματα της Αλβανίας και η Αλβανία θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί και να έχει ως πρότυπο αυτή την περίπτωση της Κροατίας. Τι θα έπρεπε να γίνεται στις, στις ε, ουσιώδεις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και μια, ένα διπλό μήνυμα σε σχέση με την Κροατία. Ναι, θέλουμε από κοινού Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο να καταφέρουμε τον Ιούνιο να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και έτσι εμείς το φθινόπωρο υπό την έγκριση που θα είναι δεδομένη να ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης. Ωστόσο όμως παρακαλούμε την Κροατία να διευθετήσει τα εκκρεμούντα θέματα, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Έχουν αναφερθεί και έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν και τα τελευταία βήματα στις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το δικαστικό και για τα θέματα των ναυπηγείων της Κροατίας. Πολλά πρέπει να γίνουν. Είναι όμως όλα αυτά πράγματα που πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να τροχοπεδίσουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να δώσουν μια δυνατότητα η Κροατία να μπορέσει να προχωρήσει και να υλοποιήσει τι υποχρεώσει. Γι' αυτό προ αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι από εδώ θα έπρεπε ένα κοινό μήνυμα να αποσταλεί προ την Κροατία αλλά και στι άλλε χώρε. Να κάνει η Κροατία σωστά το έργο της όσα πρέπει να επιτελέσει για να μπορέσει να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως αναφέρθηκε και χθε, είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθεί η Κροατία σε αυτήν όταν θα έχει επιτελέσει τα καθήκοντά της. Γι' αυτό ευχαριστούμε τους χειώδεις εισηγητές και θα πρέπει από κοινού να μπορέσουμε να αποστείλουμε αυτά τα μηνύματα προς την Κροατία και στις άλλες χώρες. Θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για την ειρηνική ολοκλήρωση της περιοχής αυτής στην Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Πόσελτ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά είμαι συγκινημένος σήμερα και το ομολογώ, διότι 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που το δημοκρατικό κίνημα στη Σλοβενία και στην Κροατία ενισχύθηκαν. Ήταν ενός έτους τότε πριν από 20 χρόνια. Υπήρξαν επεφημίες όπως και στην δημοκρατία της Τσεχίας. Μετά ήρθε όμως η ομή παρέμβαση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού τον Ιούνιο του 1990 και φάνηκε τότε ότι θα γύριζε το ρολόι πίσω και αυτό το οποίο Έλπιζε η Ευρώπη ότι θα μπορούσε να επιτελέσει μέσα στα ερήπια του Βούκοβαρ ουσιαστικά συνετρίβει. Και από τότε που ξεκίνησε η πορεία της Κροατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παρακολουθούμε και πρέπει να πούμε ότι με τεράστιες προσπάθειες ξεκίνησε και πορεύτηκε προς αυτή την οδό η Κροατία. Και ο κύριος Επίτροπος αναφέρθηκε στην αποφασιστική λέξη. Είπε ισοδίκαια πρέπει να προχωρήσουμε. Και την έκθεση Σβόμποντα θα μπορούσε να την περιγράψει κανείς ισοθή και αντιμετώπιση δικαιοσύνη προς την Κροατία. Περί αυτού πρόκειται. Όχι για εκτόσεις ή κάποια προνόμια, δίκαια αναφέρθηκε αυτό, αλλά για ισοδίκαια δικαιοσύνη, δίκαιη αντιμετώπιση. Είναι όριμη η Κροατία σήμερα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει κάποιες πρόσθετες προσπάθειες να γίνουν τους επόμενους μήνες. Όμω δεν πρέπει να δημιουργηθούν τεχνητά εμπόδια για αυτή τη χώρα όπως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γινόταν επανειλημμένα. Η Κροατία ανήκει στο ιστορικό εκείνο συνολικό πλαίσιο και στην ιστορική συγκυρία με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Θα έπρεπε με αυτές τις χώρες ως κεντροευρωπαϊκή χώρα να είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία τότε, στο παρελθόν. Λόγω πολλών άλλων γεγονότων και αιτιών δεν έγινε αυτό τότε. Τώρα όμως ορίμασε ο χρόνος και γι' αυτό πιέζουμε τώρα παραμένουμε πιστοί στη γραμμή που είχαμε χαράξει, να, είναι, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πιέζουμε όμως να μην δημιουργηθούν τεχνητά εμπόδια και αυτή η χώρα, χώρα με δικαιοσύνη ισοδίκια να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ιβο Βάιγκελ από την ομάδα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Για τελευταία φορά μιλούμε για έκθεση προόδου της Κροατίας πριν από την πλήρη ένταξη. Ο εισηγητής επί χρόνια ασχολούνταν με το θέμα της προόδου της Κροατίας και τον ευχαριστώ για την επικοδομητική του στάση. Συνεργάστηκε με όλους τους κοιόδης με άψογο τρόπο καθώς και με την κροατική κυβέρνηση. Αν εξετάσουμε τώρα υπό ποιε συνθήκες η Κροατία α, έγινε ανεξάρτητη χώρα πριν από 20 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι για πάρα πολύ χρόνο, ίσως υπερβολικά πολύ, αναμένει την ένταξη. Αναφέρετε στην έκθεσή σας όλη την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε όλοι η ένταξη να γίνει πραγματικότητα σύντομα. Πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν στο Ζάγκρεμπ. Το κεφάλαιο 23 ιδιαίτερα να προσέξουν οι φιλελεύθεροι εχθές με τον πρόεδρο Φερχόφσταντ και τον πρωθυπουργό της Κροατίας και την πρωθυπουργό της Κροατίας συζητήσαμε το θέμα της ένομης τάξης εκεί που είναι κλειδί για τον πλήρη εκδημοκρατισμό. Η διασφάλιση της ελευθεροτυπίας, της ισότητας των φύλων και της ασφάλειας για όλους είναι ουσιώδη θέματα. Και η Πρωθυπουργό ε, πρέπει να τύχει συγχαρητηρίων για τους αγώνες της σε όλους αυτούς τους τομείς. Η Κροατία εξάλλου έχει συνάψει φιλικές σχέσεις με όλες τις, τις γειτονικές πλέον χώρες. Στον τελευταίο λοιπόν γύρο των διαπραγματεύσεων και για τις τελευταίες προσπάθειες θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι όλες οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν παρόμοιες προσδοκίες και η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ένταξης όσο το δυνατόν συντομότερα γιατί μόνον έτσι θα μπορέσει η Ένωση να γίνει παγκόσμιος ηγέτης. Παρακαλώ να σέβεστε τους χρόνους σας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φραντσίσκα Κατερίνα Μπραντνερ των Πρασίνων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σπόμποντα για την καλή συνεργασία που είχαμε και πέρσι και φέτος. Είναι σωστή δίκαιη έκθεση, το είπε ο κ. Πόσελτ. Προσβλέπουμε στην σύντομη υποδοχή της Κροατίας ε, στην Ένωση. Μόλις ολοκληρώσει όλα, στηρίσει όλα τα κριτήρια, είναι σημαντική χώρα προς την ένταξη και θα είναι σημαντική ευθύνη της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι κατόπιν θα μπορέσουν και οι υπόλοιπε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν. Και από την οπτική αυτή γωνία της περιφέρειας δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τώρα είναι η καλύτερη της τάξης η κρατία, ούτως και να το πούμε αυτό, ούτως ώστε και οι λιγότερο καλοί της τάξης της να μπουν αργότερα. Θα ήταν καλό να μιλήσουμε και για τις άλλες χώρες, γιατί αν κάνουμε λάθη τώρα, πολύ πιο δύσκολο θα μπορέσουν να ε, ενταχθούν αργότερα. Αναφέρθηκε το κεφάλαιο 23 η διαφθορά. Πιστεύουμε ότι και η Ένωση θα πρέπει να εξετάσει πόσο η ίδια ενεμπλάκει σε διαδικασίες διαφθοράς και ζητούμε από την Όλαφ να εξετάσει την ευρωπαϊκή εμπλοκή στο ζήτημα. Πρέπει να είμαστε έντιμοι και έναντι του εαυτού μας. Μια τελευταία παρατήρηση. είναι σημαντικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε το παρελθόν. Ένα κομμάτι σημαντικό της ένταξης. Αναφέρθηκε το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά πιστεύουμε ότι και τα τοπικά δικαστήρια πρέπει να δουλέψουν καλύτερα. Υπήρξε μια, μια, υπήρξε μια σειρά λαθών ε, στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Είναι σημαντικό η Ένωση να υπογραμμίσει και αυτή τη διάσταση του πώς θα αντιμετωπίσει κανείς το παρελθόν του. Πάντως ε, καλωσορίζουμε, νομίζω όλοι είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε την Κροατία στην Ένωση. Ο κύριος Βαν Όντεν για τους συντηρητικούς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πιστεύουμε ότι η διεύρυνση είναι μία από τις επιτυχέστερες διαστάσεις της πολιτικής ένωσης εφόσον υπάρχουν και τηρούνται αυστηρά κριτήρια και διδαχθούμε από, τα, από τις προηγούμενες προσχωρήσεις. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία είναι κοντά. Γνωρίζουμε ωστόσο από την Επιτροπή ότι οι θέματα διαφθορά και η δικαστική μεταρρύθμιση δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και δεν είναι τεχνητέ οι ανησυχίε μα. Η Κροατία με ένα πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων ε, έχει ε, ένα backlog υποθέσεων, κάπου ένα, ε, δικαστικών υποθέσεων, κάπου ένα Ενό εκατομμυρίου. Χρειάζεται αλλαγή της νομοθεσίας για τα μέσα. Υπάρχουν υπουργοί που καταδικάστηκαν ή διώκονται για διαφθορά. Ε, δείχνουν όλα αυτά τα προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Ε, η διαφθορά στην πολιτική και τη δικαστική εξουσία δεν επέτρεψε να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα επαρκώ. Παρά τα πολλά προβλήματα ωστόσο που αναφέρονται, η, σύντομη προσχώρηση της Κροατίας είναι ε, πιθανή και θα ήταν κρίμα να γίνει η διαδικασία προσχώρησης σε ένα τυπικό στοιχείο βάσει των πολιτικών επιλογών του καθενός και χωρίς να έχουν επιληθεί τα βασικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκης Χατζηγεωργίου για την αριστερά. Ω Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, τασσόμαστε υπέρ τη ένταξη τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευελπιστούμε να γίνει σύντομα πλήρε μέλο, εφόσον αυτό είναι η θέληση του κροατικού λαού και εφόσον η χώρα εκπληρώσει όλα τα κριτήρια ένταξη. Η έκθεση προόδου και εμεί χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα τη επιστροφή των προσφύγων, στου τομεί των δικαιωμάτων των γυναικών και τη ισότητα των φύλων, καθώ και στη γεφύρωση των διαφορών με τι γειτονιάζουσε χώρε εμένουμε δε σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις ιδίως όσον αφορά τον δικαστικό τομέα και τον τομέα της πάταξης της διαφθοράς. θα πρέπει όμως να μεριμνήσουμε και για τα κοινωνικο προβλήματα που ταλανίζουν τον λαό της κροατίας όπως η φτώχεια η μακροχρόνια ανεργία η καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. δυστυχώς οι προτάσεις για προώθηση φιλελεύθερης οικονομίας θα επιβαρύνουν την κοινωνικο κατάσταση των κροατών εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε την πρόθεση μιας πραγματικά κοινωνικής ανάπτυξης που να διασφαλίζει μια ποιοτική ζωή για όλους τους πολίτες της κροατίας μέσω του εξυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας την αντιμετώπιση της ανεργίας τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες της υγείας της στέχασης, της εκπαίδευσης και της εξάλληψης των διακρίσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μειονοτικές ομάδες. ευχαριστώ.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 Πρέπει να βελτιώσουμε την τεχνική, τεχνική απόδοση. Υπάρχει πρόβλημα από τα αγγλικά και ίσως και σε κάποιες άλλες καμπίνες. Όχι ακόμα, δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Πρέπει κάτι να βελτιώσουμε. Yes, please, start. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Μικροφωνίζει πάλι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ένα τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Οι τεχνικές υπηρεσίες θα επιληφθούν άμεσα. Uh, Συνάδελφε Πάσκα, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή εκφωνώντας τον λόγο σας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Μικροφωνίζει πάλι, δυστυχώς. Ε, Μικροφωνισμός. Ε. I'm very, very sorry. Something really Κύριε Πάσκα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο μικροφωνισμό. Το πρόβλημα είναι στα αγγλικά ή σε όλες τις γλώσσες, λέει ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσουν να την οροπήσουν οι τεχνικοί μας. Μου ζητήθηκε να μιλήσω πολωνικά για να δούμε αν η αγγλική διερμηνία λειτουργεί. Γιατί όταν μιλάω στα αγγλικά δεν μπορώ να, μιλ... να... να ελέγξουμε. Λοιπόν, έχουμε παρακαλώ, ζητώ κάποια λίγα λεπτά χρόνο και υπομονή. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λειτουργεί λοιπόν. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, συνάδελφε Πάσκα, παρακαλώ τον κύριο Πάσκα να ξεκινήσει το λόγο του και πάλι. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Κύριε... Κύριε Υπουργέ, από τον Οκτώβριο 2005, όταν είχε τότε ληφθεί η απόφαση για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τελικό στόχο φυσικά αυτή την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Η τελευταία πιο σημαντική πρόοδος έγινε το 2010 όταν κατάφερε η Κροατία και ολοκλήρωσε διαπραγματεύσεις σε αρκετά περίπλοκα κεφάλαια και επίσης έκανε και σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές του συντάγματός της και συνέχισε να βελτιώνει τις σχέσεις της ε, στα σύνορα με γειτονικέ χώρες ε, και σε σχέση με επίσκεψη που έγινε στο Βουκόβαρα καταδείχθηκε ότι οι σχέσεις Κροατών και Σέρβων μπορούν να οικοδομηθούν με βάση την αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαίο σεβασμό. Γι' αυτό η ταχύτητα και ο ρυθμός ε, ολοκλήρωσης ε, βρίσκεται πλέον στα χέρια των Κροατών των ιδίων αυτή τη στιγμή. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το έργο τους στην διαδικασία της ολοκλήρωσης ε, των κεφαλαίων που εκκρεμούν ακόμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρος. Στη συνέχεια σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος αγωνιτής, ε, ο κύριος Ανδρουθόλ, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από 20 χρόνια η Κροατία αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία τη. Τώρα την παραδίδει χωρί ούτε μια σφαίρα. Υποχρεούται να κάνει σημαντικέ νομοθετικέ αλλαγέ ε, και να αποστείλει την υποστήριξη από μια σειρά βιομηχανικών κλάδων. Για... Και όλα αυτά για να δεχτεί η, η Ένωση την Κροατία. Επιπλέον όλες αυτές οι αλλαγές παραχωρούνται χωρίς να υπάρξει συνένεση των πολιτών ε, μέσω δημοψηφίσματος. Ουσικά καν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Παρά τις φυγμομετρήσεις ότι η πλειοψηφία είναι κατά της ένταξης στην Ένωση, θεωρείται ως δεδομένο ότι το δημοψήφισμα θα είναι θετικό οι τεράστιες αυτές αλλαγές εν ώψη των λαμβάνουν χώρα χωρίς της, τη συνένεση. Οπότε θεωρεί, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι τυπικό μόνο το OK των πολιτών. Η έκθεση εδώ αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι ε, διαμαρτύρονται για πολιτικές πιέσεις αλλά κανείς δεν μιλά για την παρεμπόδιση της ελεύθερης εξαγωγής του δημοψηφίσματος. Ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητές. Ο κ. Σέλμαρ Μπρόκ, ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά βρισκόμαστε στο τελευταίο γύρο τώρα, στην τελευταία ευθεία, πριν από την ένταξη της Κροατίας ε, εφόσον ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του. Διότι θα έχουμε και την καθόλου απλή στη συνέχεια διαδικασία επικύρωσης μια και παρακολουθήσαμε και τις προηγούμενες διευρύνσεις με τα προηγούμενα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παρακολούθησα του σύνεγγυς ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και αναφέρεται ότι η Κροατία είναι μια χώρα που σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκε για την υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός ο γύρος θα στεφθεί με ένα ναι αυτή θα είναι η τελική έκβαση. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ένα μήνυμα προς τις άλλες πολλές χώρες που αναμένουν να δουν ότι η θύρα προς την Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και δεν έχει κλείσει. Και κάτι άλλο το οποίο ισχύει ακόμα. Με βάση την πείρα μας με άλλες χώρες πρέπει να πούμε ότι η Κροατία προς το ίδιο συμφέρον της, άσχετα από τη διαδικασία της ένταξης, πρέπει να προχωρήσει για την μεταρρύθμιση στο δικαστικό ε, σκέλος, για παράδειγμα. Υπάρχουν ε, κατηγορίες που εγείρονται για θέματα διαφθοράς, ε, οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και όλα αυτά είναι, υπονομεύουν τη συνολική εξέλιξη αυτής της χώρας. Ευχαριστώ. Επόμενο αγορητής. Ο κύριος Γιώραν Φάρμα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Σφόμποντα για την έκθεσή του. Εξαιρετική δουλειά. Η προσχώρηση της Κορατίας έρχεται όλο και πιο κοντά. Λίγα ζητήματα που αφορούν την διαφθορά παραμένουν εκκρεμή. Βελτίωσε η κορατία την νομοθεσία της, ωστόσο τώρα πρέπει να την υλοποιήσει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την δικαστική ανεξαρτησία. Είδαμε τον κύριο Σαναντέρ και μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το θάρρος των δημοσιογράφων που ε, αναφέρθηκαν στην διαφθορά. Η διαφθορά βέβαια προέρχεται από όλες τις πλευρές ε, υπάρχουν καταγγελίες ότι ο κύριος Ανδρέα προσπάθησε να επηρεάσει με, εσφαλ, με, ανάρμοστο τρόπο την Ένωση και θα πρέπει η Όλαφ να ελέγξει απόλυτα και να διαφωτίσει το τι έγινε στο παρελθόν. Θέλει το ΕΛΚ να διαγραφεί το, τμήμα αυτό ε, του ψηφίσματος, ωστόσο πρέπει να είμαστε ε, και διενεργοί, να μην ε, αφήνουμε τα πράγματα στην άκρη. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην φάση, σε μια φάση κρίσης είναι καλό να βλέπουμε ότι η Κροατία προχωρά προς την ε, προσχώρηση. Σημαντική πρόοδο πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να, να μας οδηγήσει στο να γνωρίσουμε ότι πολλά πράγματα παραμένουν να γίνουν ακόμα. Δύο θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ. Ενίσχυση του, της δικαστικής εξουσίας. Μια ισχυρή δικαστική και ανεξάρτητη δικαστική εξουσία είναι αναγκαία για να, για να καταπολεμηθεί η διαφθορά, για να υπάρξει μακροπρόθεσμα κράτος δικαίου. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίζουμε τους ε, εγκληματίες μόνο, αλλά και να τους προλαμβάνουμε. Η δεύτερη, ε, δεύτερο θέμα, η ανάγκη να υπάρξει στην κοινωνία μια κοινωνία, στην Κορατία μια κοινωνία ανεκτικότητας που θα στηρίζεται στη συμφιλίωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο χώρε. Εγώ χαιρετίζω την βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονε τη Κροατίας. Αλλά πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση και στο εσωτερικό της χώρας. Οι απειλέ βίας κατά το μειονοτήτων είναι απαράδεκτες. Κατανοώ πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι και οι διαπραγματεύσει και οι συνέπειες της διεύρυνσης θα είναι θετικές για την ε, κοινωνία της Κροατίας. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή ε, θα λάβει τον λόγο παρακαλώ ο κύριο ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χωρί καμία αμφιβολία θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Κροατία να επιτελέσει του φιλόδοξου στόχου τη Πρόκειται για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ένταξη τη Κροατία στην Ένωση μέχρι τα τέλη αυτού του πρώτου εξαμήνου του 2011. Μα δίνει μια σημαντική χώρα ω εταίρο και σύμμαχο η δυνατότητα αυτή για τη σταθεροποίηση τη περιοχή και ένα υπόδειγμα για πολλέ άλλε χώρε των Βαλκανίων που ενδιαφέρονται και εκείνε για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό μου με κάθε τρόπο για τις μεταρρυθμίσεις ε, που έχει επιτελέσει η ε, κυβέρνηση της Κροατίας, ιδιαίτερα στον τομέα, στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς, ε, του οργανωμένου εγκλήματος κτλ. Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα και υπάρχουν προβλήματα τα οποία ακόμα πρέπει να επιληθούν. Εύχομαι να γίνει αυτό το δυνατόν ταχύτερα. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες από την ίδια την Κροατία που μας λένε και δείχνουν ότι οι Κροάτες δεν έχουν πιστεί 100% απόλυτα ότι θα είναι θετική η ιδιότητα κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα τους. Τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να αναλυφθούν ώστε να αναχαιτιστεί αυτή η τάση. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο εσείς για ένα λεπτό κύριε Βέλγερ παρακαλώ. Ο κύριος Μπέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει σημειώσει, έχει επιτελέσει θετικές πρόοδους ε, η Κροατία καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι διαμφισβήτο και με ικανοποιεί. Υπάρχει όμως ένα σημείο για το οποίο ανησυχώ. Η διαφθορά σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων έχει μεγάλες διαστάσεις και βλέπουμε στα εδάφια 7 και 8 της πρότασης ψηφίσματος τη σχετική διατύπωση. Αυτό επηρεάζει και την οικονομία και τις εμπορικές μας σχέσεις με τη χώρα αυτή. Χρειάζεται μια καλύτερη, πιο θετική προσέγγιση για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. Τότε βλέπουμε ότι και στην παράγραφο 28 υπάρχει και ένα άλλο κακό κείμενο, δηλαδή κακές διοικητικέ πρακτικές. Χρειάζεται μια σωστή διοικητική μεταρρύθμιση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι της Κροατίας. Εφόσον δεν έχουν επιληθεί αυτά τα δύο προβλήματα τα οποία προανέφερα, ανησυχώ πρέπει να πω. Ανησυχώ δεδομένη τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου προτίθεται να ε, ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει με την Κροατία. Θα έλεγα η ίδια η ένταξη της Κροατίας δεν αμφισβητείται. Η ποιότητα όμως της ένταξής της είναι σημαντική και είναι σημαντικό για την αποδοχή των Ολλανδών αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ κυρία Αγγέλικα Βέτμαν παρακαλώ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνολικά οι εξελίξεις στην Κροατία βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Η θεωρία έχει υλοποιηθεί πλήρως, στην πρακτική εφαρμογή πρέπει να γίνουν πολλά. Τρία πράγματα εκκρεμούν ακόμα και πρέπει να επιτελεστούν. Πρώτον, η Κροατία πρέπει πιο έντονα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να συνεργαστεί στη Χάγη, ώστε το θέμα της δίωξης των πρώην εγκληματιών πολέμου να προαχθεί και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει wall of silence. Υπάρχουν σημαντικές περιπτώσεις ε, περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα ήταν πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε συμβιβασμού σε αυτό. Δεύτερον, το θέμα της διαφθοράς. Αυτό το θέμα διαποτίζει την κοινωνία και την πολιτική στην Κροατία. Χαιρετίζουμε τι προσπάθειε τη Κροατία να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην ίδια τη χώρα αυτή. Ταυτόχρονα πρέπει να πιέσουμε όμω αυτό το πρόβλημα να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με μεγάλο σθένο. Τρίτον, η Κροατία πρέπει προ το ίδιο συμφέρον τη χώρα να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσει που έχουν ξεκινήσει, για παράδειγμα στη δικαιοσύνη, θα συνεχιστούν με ταχύ ρυθμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λίσεκ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι. Όταν πριν από δύο χρόνια βρισκόμουν ακόμα στο Πολωνικό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και υποδεχθήκαμε συναδέλφους από την Κροατία, αυτοί οι συνάδελφοι μου έθεσαν το εξής ερώτημα. Γνωρίζετε, είπαν, πόσοι ιστιοπλόοι από την Πολωνία τώρα ασχολούνται με το άθλημά του στην Κροατία. Χιλιάδες είναι, χιλιάδες, είναι εκατομμύρια τουρίστες που πάνε κάθε χρόνο σε αυτή την υπέροχη χώρα και είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι αυτή η χώρα, δηλαδή η Κροατία, είναι έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι συνάδελφοι έθεσαν το ερώτημα πώς αντιμετωπίζει η Πολωνία το θέμα της αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων της. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτά που ανέφερε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου κύριος Μάρτονη θα γίνουν πραγματικότητα. Εκινούμε από το ότι η Προεδρία θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και θα ακούσουμε και από τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας σηκώσει ότι συνεχίζονται αυτές οι προσπάθειες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σφόβοντα για το έργο του. Σε ό,τι αφορά την Κροατία, θα ήθελα πραγματικά να είναι η τελευταία έκθεση και να προσχωρήσει η Κροατία στην Ένωση το συντομότερο δυνατό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει η Κροατία να προλάβει τις ε, καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπτυξη των πολιτισμών, της οικονομίας, των, του, του πολιτισμού, της οικονομίας των τεχνών, η Κροατία ήταν πάντα ε, μαζί στην ίδια κατηγορία με τις χώρες που μπήκαν πριν από χρόνια στην Ένωση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις αρχές του Ζάγκρεμπ, διότι έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να καταπολεμήσουν την διαφθορά. Η προστασία των δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης είναι κάτι που επίσης πρέπει να προσέξουμε. Η ένταξη της Κροατίας στην Ένωση σημαίνει ότι προσφέρουμε μια χείρα βοηθείας και προς τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια. Προσβλέπω λοιπόν να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους για την ειρήνη στην περιοχή. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Σβόμποντα για την καλή δουλειά που έχει κάνει και ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία έκθεση πριν υπογράψει συνθήκη Προσχώρηση η Κροατία. Πιστεύω ότι η ένταξη της Κροατίας στην Ένωση θα αποτελέσει ε, μια παρότρινση για την ειρήνη στην περιοχή. Το έδειξε αυτό η Κροατία μόνη της παρέχοντας ε, χωρίς ε, να υποχρεωθεί μεταφράσεις πολλών σελίδων του κεκτημένου της Ένωσης στους γείτονές της, δείχνοντας έτσι ότι μπορεί να συμβάλλει, είναι πρόθυμη να συμβάλλει στην προσχώρηση ολόκληρης της περιοχής στην Ένωση. Παρότι κάθε χώρα στην Ήπειρό μας έχει τα προβλήματά της, δεν θα έπρεπε να δείχνουμε με το δάχτυλο τις ανατολικές χώρες μόνο όταν μιλούμε για διαφορά και για προβλήματα στη δικαστική εξουσία. Δεν είναι χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής μόνο με συνεργασία μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Η διαφάνεια είναι, βασι... είναι αρχή και θα έπρεπε να παροτρύνουμε τα Δυτικά Βαλκάνια να το αντιμετωπίσουν. Καλή επιτυχία στην Σλοβακία. Στην Κροατία, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνει τα πράγματα όπως πρέπει διότι όταν μπήκαν πριν από έξι χρόνια οι καινούργιες χώρες ήδη είχαν φανεί οι φραγμοί για την ένταξη της Κροατίας. Έκτοτε είχαμε πει ότι είναι προτεραιότητα η ένταξη αυτή. Η ενοποίηση της Ευρώπης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τις χώρες των δυτικών λεγόμενων Βαλκανίων. Όλες οι χώρες της πρώην Νοτιοσλαβίας είναι εκτός ένωση, εκτός από τη Σλοβενία. Και πρέπει η κατάσταση αυτή να αλλάξει. Αν ενταχθεί φέτος η Κροατία θα γίνει ένα τεράστιο βήμα προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Έχουμε ηθικό καθήκον να ενθαρρύνουμε τις χώρες αυτές της Ευρώπης γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. 18 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Καταλαβαίνετε δεν μπορούν να πάρουν το λόγο όλοι διότι η διαδικασία περιλαμβάνει μόνο χρόνο πέντε λεπτών. Ε, πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πολλοί συνάδελφοι θέλουν να εκφραστούν, οπότε θα πάρουν το λόγο μόνο έξι συνάδελφοι και σας παρακαλώ για ένα λεπτό ο καθένας. Ε, θα και θα προσπαθήσω να κρατήσω τη σειρά ε, βάσει της προτεραιότητας που έχουν οι συνάδελφοι αφόσον ζήτησαν το χρόνο. Ο κύριος Έρτζιμπ θα πάρει το λόγο πρώτος για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και η έκθεση, έκθεση Σβόμποντα, αλλά και η έκθεση της ίδιας της Προεδρίας και τα όσα ακούσαμε από τον Επίτροπο Φίλε δείχνουν ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα, μια πολύ καλή ατμόσφαιρα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει επίσης να τονίσουμε και την βούληση της ίδιας της Κροατίας που είναι δεδομένη να μπορέσουν να ολοκληρωθούν ταχαίως οι διαπραγματεύσεις αυτές και να συνεργαστεί η Κροατία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Αυτή η προοπτική λοιπόν ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και το θετικό κλίμα, η θετική ατμόσφαιρα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν την Κροατία την ίδια που αναμένει 20 ολόκληρα χρόνια και που τώρα θα ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος αναμονής με την ολοκλήρωση της συνθήκης, υπογραφή της συνθήκης συμβολικά και πρέπει να τιμηθεί αυτή η προσπάθεια διότι η Κροατία σε όλες τις γειτονικές χώρες διέθεσε μεταφρασμένα τα κείμενα για τα κεφάλαια της ένταξης. Υποθέτω ότι η έκθεση Σβόμποντα θα είναι η τελευταία για την πρόοδο της Κροατίας και θα χαιρετήσουμε την Κροατία σύντομα ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα μπάτσι θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Τίστερ Μπίστος úr, miniszter úr, egyértelműen támogatom. Πρόεδρε, επίτροπε, κύριε Υπουργέ, Συμμερίζομαι απόλυτα τις ε, προσπάθειες της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του εξαμήνου η διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Η ε, χώρα υποχρεούται να κάνει αλλαγές σημαντικότερες από αυτές μερικές φορές των κρατών μελών, πρέπει να καλυφθούν ε, μια σειρά κεφαλαίων που ανέφερε και ο Υπουργός ε, τα υπογράμμισε σωστά ο κύριος Φόμποντα. Οι δυνατότητες ε, της ε, η ένταξη της Κροατίας θα προσφέρει προοπτικές και για άλλες περιοχές της ε, και για άλλες χώρες της περιοχής, Σερβία για παράδειγμα, προς το συμφέρον όχι μόνο της Ένωσης αλλά και των λαών. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι αλλαγές είναι βασικές για αυτούς. Είναι αναγκαίο να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης των μειονοτήτων στην περιοχή, ιδιαίτερα των Σέρβων στην Κράινα, να καταλάβουμε και την κατάσταση αλλά και την κατάλαβη την κατάσταση της κοινωνίας. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε τις χειρονομίες που έκανε και ο αρχηγός του κράτους της Κροατίας προς την Σερβία και την υπόλοιπη περιοχή. Γιατί θα έχουμε τις ψηφοφορίες στις 12. Ο κύριος Κατσίν έχει το λόγο τώρα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ελπίζω και η Κροατική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξουν την απαραίτητη επιμονή και ενέργεια ώστε ίσως η, στην επέτειο της ε, ανεξαρτησίας της Κροατίας να γιορτάσουμε και την ένταξη. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τη σταθερότητα και συνεργασιμότητα της κυβέρνησης της. Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι μεγαλύτερη ευαισθησία των πολιτικών. Η σοβαρή οικονομική κρίση μειώνει τα ωφέλη που βλέπουν οι πολίτες σε πολύ χαμηλά περιθώρια και οι διαπραγματεύσεις δεν θα έχουν μεν καταστροφικές επιπτώσεις για την Κροατία αλλά μπορεί να δοθεί ένα πολύ αρνητικό μήνυμα για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ζητούν και αυτές την ένταξή τους. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις θα απογοητευτούν όλοι, να το ξέρετε. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πρέπει να πω ότι η Κροατία πλησιάζει, προσεγγίζει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο προϊονίζονται θετικά και η ένταξη άλλων χωρών και της ε, Τουρκίας μελλοντικά. Αλλά είμαστε τόσο πολύ υπέρ, εμείς, ε, υπέρ της Κροατίας επειδή οι μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθεί η ένταξη είναι τόσο σημαντικές. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα η Κροατία. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αναφέρεται κάποια ημερομηνία στην έκθεση. Ίσως θα μπορούσαν οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011. Ίσως και όμως όχι. Δεν είναι σημαντικό πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Σημαντικό είναι η Κροατία κατά τη χρονική στιγμή που, της ένταξης να υλοποιεί όλα τα κριτήρια. Αν μάθαμε κάτι από την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι ακριβώς αυτό. Να μην αναφέρετε κάποια ημερομηνία αλλά να αναφέρετε τι πρέπει να έχει επιτευχθεί πιο πριν, πριν από την ένταξη. Και ένα σημείο στο οποίο μπορεί να κάνει κάτι η Κροατία είναι η, προστασία των μειονοτήτων. Ωραίο θα ήταν αν η από πλευράς ε, της Προεδρίας θα μπορούσε να δοθεί ένα καλό παράδειγμα η Βουδαπέστη να ακολουθούσε αυτές τις αρχές η ίδια καλύτερα ευχαριστώ. Όπως αναφέρει η έκθεση προχωρά σημαντικά. Εμεί υποστηρίζουμε την Κροατία στην τήρηση των κριτηρίων τη Κοπεχάγη. Η, Ευρω... μεγαλύτερη, η ευρύτερη ένωση θα είναι πιο ευέλικτη και λιγότερο συγκεντρωτική. Η Κροατία θα έπρεπε να επενεθεί για τι προσπάθειε να αντιμετωπίσει την διαφθορά όπω ε, και την δίωξη του κ. Σαναντεχέρο που η Σλοβενία δεν μπλοκάρει πλέον την προσχώρηση τη Κροατία. Ήταν ένα διμερέ θέμα αυτό και το οποίο δεν θα έπρεπε να εμποδίσει την ένταξη τη Κροατία στην Ένωση. Ε, και το, η μικρή διαφθο, για διαφορά, συνολική διαφορά που έχει με το Ευρωβούνι ε, πρέπει να λυθεί μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να βοηθήσει τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων ως εισηγητής για το Μαυροβούνι. Θα ήθελα να ζήσω και από το Μαυροβούνι και την, και την Σερβία να προχωρήσουν τις ε, μεταρρυθμίσεις και να μην μπλοκάρει η Κροατία την ένταξη της Σερβίας. Ένα λεπτό παρακαλώ θα πάρει το λόγο. Ε, Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ των υποψήφιων για ένταξη είναι γνωστό ότι η Κροατία έχει τις μεγαλύτερες πρόοδους που σημειώνει για την ένταξη και αυτό δεν μας εκπλήσει. Η Κροατία επανειλημμένα απέδειξε την ικανότητά της καθώς επίσης και για την διευθέτηση του προβλήματος αλληλείας με τη Σλοβενία. Φυσικά υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν, όμως ε, είναι δεδομένη ε, η, θέληση και η βούληση της ε, Κροατίας να ολοκληρώσει. Σε σχέση με τους εγκληματίες πολέμου αρκετά έχουν κινητοποιηθεί τα πράγματα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με πρώην υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών. Και πρέπει να δούμε και σε σχέση με την υποστήριξη για την επιστροφή των προσφύγων τι μπορεί να γίνει. Σημαντικό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδιαφέρεται όχι μόνο για την επιστροφή των εκτοπισμένων αλλά και για την επιστροφή των προσφύγων και σημαντικό για τη θέση των ε, Σουηβών εκεί. Ευχαριστώ. Κύριο Σοντή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω την ισορροπημένη έκθεση του συναδέλφου Σβόμποντα. Πρέπει η ένταξη αυτή να επιτευχθεί οπωσδήποτε. Και αυτό με οδηγεί στο να σχολιάσω τι μεγάλες και σοβαρές αντιρρήσεις που βλέπουμε στην κοινή γνώμη να σημειώνονται για την ένταξη αυτή. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου έγινε μια ολόκληρη σειρά εντάξεων πρώην κομμουνιστικών χωρών και σήμερα κυρία Επίτροπε νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει μια μεγάλη καμπάνια πληροφόρησης, επικοινωνία σε όλες τις χώρες και ίσως και στην Κροατία για να εξηγηθεί όλη η εργασία που, η προεργασία που έγινε ώστε να εξηγηθεί ότι η ένταξη αυτή έχει προετοιμαστεί σωστά. Αυτό προτείνω διότι η ένταξη δεν είναι ενωσιακή δικαιοδοσία αλλά εθνική και πρέπει να την πετύχουμε να μην αφήσουμε κανένα μέσο ανεκμετάλλευτο για να επιτύχει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Τελειώσαν εδώ οι παρεμβάσεις δυστυχώς των συναδέλφων και το, ρόλο, ε, το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος, ο κύριος Φούλε. Mr. Commissioner. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θέλω καταρχά να σα ευχαριστήσω για την επικοδημητική και ενθαρρυντική συζήτηση. Το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου με το ισορροπημένο μήνυμά του είναι ζωτική σημασίας για την Επιτροπή προσφέροντας ε, σημαντικές πληροφορίες και κατευθυντικές γραμμές για την ε, τις διαπραγματεύσεις ε, με την Κροατία. Έγιναν πολλές φορές ε, αναφορές για την ε, ευθυδική ποιότητα και ακρίβεια της, της έκθεσης αυτής. Πολλές από τις παρεμβάσεις σήμερα υπογράμμισαν ότι χρειάζονται πολλές ακόμα προσπάθειες οι οποίες όμως είναι προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Αυτά τα ωφέλη πρέπει να περάσουν σαφώς στον ε, πληθυσμό τους επόμενους μήνες. Κυρίε και κύριοι, η υποστήριξη, η στέρεη υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην ενταξιακή διαδικασία τη Κροατία είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Σημαντικό όχι μόνο για την Κροατία, αλλά για όλε τι υποψήφιε και εν δυνάμει υποψήφιε χώρε. Η υποστήριξή σα, μάλιστα, θα του ενθαρρύνει, θα ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να συνεχίσουν εντατικά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης των παρελθών και θα βοηθήσουν την ταχύ ολοκλήρωση των ενταξιωκών διαπραγματεύσεων. Στου Συμβουλίου θα πάρει λόγο τώρα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εξ ονόματος της Προεδρίας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για την δουλειά του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα του εισηγητού σας Χάνς Σβόμποντα που συνεχώς και αδιαλείπτος έκανε την προσπάθεια όχι μόνο για να πετύχει η ένταξη της Κροατίας αλλά και για να προοδεύσει γενικά η διαδικασία της διεύρυνσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες φαίνονται από την τη σημερινή συζήτηση. Επίσης πιστεύω ότι το ψήφισμα που θα εγκριθεί θα τονίζει τον ζωτικό, θα δείχνει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων και για την ένταξη της Κροατίας. Δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, στους πολίτες της Ευρώπης, ότι πράγματι δηλαδή η διεύρυνση εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και θα τους πείσει ότι ίσως η κούραση που έχουν επιδείξει για τις διευρύνσεις, αζαβλεπάλες διευρύνσεις, έχει υποχωρήσει μπροστά στο στόχο της Ένωσης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως θα είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα και για τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Το λέει το ψηφισμά σας βεβαίως και όλοι γνωρίζουμε ότι ο παράγων κλειδί της σταθερότητος, της συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι το ευρωπαϊκό όραμα και η προοπτική που πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη και να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα και απτά μέτρα όπως ακριβώς η επικείμενη ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκκρεμή θέματα, η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο βασικός μας στόχος είναι η διαδικασία αυτή να συνεχίσει. Ορισμένα σημαντικά σχόλια ακούστηκαν παραδείγματος χάριν Πράγματι εδώ και έξι χρόνια συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις, ήταν μακρά η διαδικασία μακρύτερη από ό,τι από άλλες χώρες. Τώρα όμως πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να επιταχύνουμε τη διαδικασία όσο μπορούμε. Πολλές επιτεύξεις έχουν σημειωθεί και από τις δύο πλευρές, πολλά επιτεύγματα και πρέπει να ξανατονίσουμε την θέλησή μας να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να υπάρξει μια καλής ποιότητας διεύρυνση. Αυτό το μήνυμα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας και μέσα και έξω από την τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για τα σημαντικά σας σχόλια και εκφράζω τις ευχαριστίες μου και προς την Κομισιόν. Ελπίζουμε να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε τους στόχους μας και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις πριν λήξει ο χρόνος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την ε, συζήτηση αυτή, για το θέμα της συζήτησης αυτής. Έληξε η συζήτησή μας και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα δηλαδή. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι κοινή συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη 2020, κατευθυντήριε γραμμέ για την πολιτική απασχόληση. Έχουμε τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε την έκθεση μπέρε. Ε, που